Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας κύριε Ναπολετάνο. Ε, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και χαρά που σας ε, υποδεχόμαστε στην συνεδρίασή μας. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλώς ήρθατε σε αυτή την έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών που ασχολείται εκτός από τις πολιτικές ελευθερίες με τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις και έχουμε μαζί μας φυσικά και την μεικτή κοινοβουλευτική αντιπροσωπεία σχέσεων με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Είναι μια μεικτή έκτακτη συνεδρίαση δηλαδή. Ο κύριος Έλμαρ Μπρόκ είναι ο πρόεδρος αυτής της κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας και αυτό συμπροεδρεύουμε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση. Έχουμε μια μοναδική ευκαιρία για την ενίσχυση του διατλαντικού διαλόγου με την ενεργό συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το να εκλεγέν αυτό κοινοβούλιο βρίσκεται μπροστά σε πολλές αλλαγές, γιατί επιτέλους θα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας από την 1η Δεκεμβρίου, κάτι που σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενδυναμωθεί περισσότερο από ποτέ. Το κοινοβούλιο αυτό θα πλέψει ολοταχώς για να αναπτύξει κοινοβουλευτική διπλωματία και θα έχει αποφασιστικό ρόλο στις αποφάσεις για νομοθετικά ζητήματα. Για ζητήματα που μέχρι στιγμής ανήκαν στον τρίτο πυλώνα και τη δια κυβερνητική συνεργασία. Τώρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα έχει το λόγο του σε θέματα δικαιωμάτων, ηθαγένειας, εξωτερικών συνόρων, μετανάστευσης, ασύλου, δικαστική συνεργασία για ποινικά και πολιτικά ε, και αστικά ζητήματα, καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, της λεύκασης, η νομοποίηση παράνομου χρήματος, τρομοκρατία. Όλες αυτές οι απειλές ε, είναι πραγματικές και στην Επιτροπή μας αλλά και σύσσωμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι προσιλωμένο στο στόχο γι' αυτό και καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά ε, την ε, νέα κυβέρνηση Ομπάμα που μόλις συμπλήρωσε ένα χρόνο θητείας και φυσικά καλωσορίζουμε και τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών με επικεφαλή στην Υπουργό Ναπολετάνο. Η κυρία Ναπολετάνο γνωρίζει τα πράγματα εκ των έσω, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την πρόσφατη επίσκεψη της κοινοβουλευτικής μας αντιπροσωπείας στις Ηνωμένε Πολιτείες. Βρεθήκαμε εκεί επ' ευκαιρία της ε, υπογραφής ενός πολύ σημαντικού πακέτου συμφωνιών κυρίως μιας διμερούς συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών για την αμοιβαία νομική αρρωγή και μια άλλη διμερή συμφωνία για τις εκδόσεις. Μάλιστα η κυρία Ναπολετάνο ήταν πρόσφατα στη Μαδρίτη και έλαβε μέρος σε μια σημαντική παγκόσμια διάσκεψη για την προστασία των δεδομένων. Και είναι και αυτή προσιλωμένη στο στόχο ανέβρεση νέα ισορροπία μεταξύ τη ελευθερία, τη ιδιωτική σφαίρα αλλά και τη ασφάλεια. Γιατί αυτή είναι η προτεραιότητά μα και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλά από τα θέματα αυτά ε, συζητήθηκαν πρόσφατα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Γιατί είχαμε τις ε, εκθέσεις για το PNR και το SWIFT. Οπότε η κυρία Ναπολετάνο γνωρίζει ότι η Επιτροπή μας απασχολείται με τέτοια θέματα, είναι πολύ δραστήρια Επιτροπή και η ευκαιρία αυτή είναι πολύ σημαντική. Και η κυρία Ναπολετάνο ε, είναι υπέρ ε, σύσφυξης των σχέσεων και του διαλόγου μεταξύ μας. Έχουμε μία ώρα και κάτι και αυτή η ευκαιρία πραγματικά θα είναι πολύ χρήσιμη γιατί θα δείξει την προθυμία μας ε, για συνεργασία και ενεργό διάλογο με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη, το σεβασμό, την αποφασιστικότητα, αλλά φυσικά και την αμοιβαιότητα. Γι' αυτό, κύριε Υπουργέ, κύριε Ναπολετάνο, καλωσορίσατε και πάλι και έχετε το λόγο. thank you very much and, uh, thank you. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να έρθω εδώ σε αυτή την έκτακτη συνάντηση. Είναι πολύ επίκαιρη η στιγμή και νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα επικοδομητικό διάλογο. Εκπροσωπώ την κυβέρνηση Ομπάμα και έρχομαι εδώ με την αίσθηση ότι έχουμε κοινέ αξίες όπου η ιδιωτική σφαίρα και η ασφάλεια μας απασχολούν και από κοινού προσπαθούμε να φτάσουμε σε μια κοινή ευρεία συμφωνία για το πώς θα μοιραζόμαστε τις πληροφορίες. Πιστεύω ότι μια κοινή συνεργασία για θέματα εγκλημάτων και τρομοκρατίας που δυστυχώς ε, δεν έχουν φραγμούς και που είναι στοιχεία του περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργούμε, είναι απειλές το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε. Εμείς είμαστε εδώ λοιπόν για να μειώσουμε τον κίνδυνο. Νομίζω ότι προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα με αμοιβαίο σεβασμό. Βεβαίως ε, ερχόμαστε εδώ ε, με διαφορετικές παραδόσεις, διαφορετικές κουλτούρες, αλλά κοινού στόχους και το πώς θα υλοποιήσουμε αυτούς τους στόχους είναι ακριβώς η πρόκληση που αντιμετωπίζουμε στο εγγύς μέλλον. Χαίρομαι λοιπόν για αυτή τη συνάντηση σήμερα, για τη δυνατότητα να συνδιαλλαγούμε, να ακούσω τις ερωτήσεις σας για κάποια από τα θέματα που μας απασχολούν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία και για το ότι οργανώσατε αυτή τη συνάντηση. Πολύ ωραία. Ας περάσουμε στην ουσία και στις ερωτήσεις. Βλέπω ότι διάφοροι ζήτησαν τον λόγο. Ο κύριος Κάρλος Κοέγιο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω την Υπουργό Νεπολετάνο αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά και τιμή και προνόμιο που βρισκόμαστε σε αυτή την κοινή συνεδρίαση και χαίρομαι που θα ακούσετε και τη φωνή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε να τροφοδοτηθεί ο διάλογος και να εξασφαλιστεί αυτή η αμοιβαιότητα που είναι πολύ σημαντική. Σας λέω ειλικρινά ότι έχουμε υψηλές προσδοκίες από την κυβέρνηση Ομπάμα Δυστυχώ, οι σχέσεις ε, Ηνωμένων Πολιτειών Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν βρέθηκαν ε, στην καλύτερη του στιγμή με την προηγούμενη κυβέρνηση. Με την κυβέρνηση Bush είχαμε πολλά προβλήματα. Τα συζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είχαμε την περίπτωση SWIFT και τον τρόπο που εφαρμόστηκε το PNR. Επίσης υπήρξε ένα διχασμός μεταξύ των χωρών τη παλιά και τη Νέα Ευρώπη. Θυμόμαστε τι δηλώσει του Ράμσφελτ και τη διάκριση που έκαναν οι Αμερικανοί μεταξύ των παλιών και νέων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης είχαμε παράνομες δραστηριότητες CIA στην Ευρώπη γι' αυτό και συστήσαμε ειδική εξεταστική επιτροπή και είχαμε και την περίπτωση του Γουαντάναμου. Όπως ξέρετε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ζήτησαν ε, κατηγορηματικά το κλείσιμο του Γουαντάναμου και αισθανθήκαμε ιδιαίτερη χαρά με τη σχετική απόφαση του Πρόεδρου Ομπάμα και είπε κάτι που μας άγγιξε πραγματικά, ότι θα πρέπει να, ανακτήσει οι να ανακτήσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, το κύρος και την ηθική τους αυθεντία. Γιατί αυτό χρειαζόμαστε, μια ε, Αμερική, Αμερική, Ηνωμένε Πολιτείε που να σέβονται τον νόμο, που να σέβονται τις ηθικές αρχές και δεν θα παραβιάζουν επουδενή ε, στο βωμό της καταπολέμησης του εγκλήματος της πολιτικές ελευθερίες. Θέλουμε λοιπόν αμοιβαιότητα στο σεβασμό του διεθνούς και εθνικού δικαίου και σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ε, για τα θέματα αυτά. Έχω δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις. Το θέμα της διαφάνειας και της πρόσβασης στα έγγραφα. Στο παρελθόν, όταν είχαμε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, το Συμβούλιο της Ένωσης αρνήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, την πρόσβαση στα έγγραφα. Ε, ζητώντας, ε, με το πρόσχημα ότι αυτό ήταν το αίτημα των Αμερικανικών αρχών. Ελπίζω ο Ομπάμα να μην κάνει το ίδιο με την κυβέρνηση Μπούς. Δηλαδή να μην ζητήσει η κυβέρνηση Ομπάμα να παρεμποδιστεί η πρόσβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα δημόσια έγγραφα των συζητήσεων μεταξύ Συμβουλίου και Ηνωμένων Πολιτειών. Σε ό,τι αφορά την υπογραφή των συμφωνιών, της Ουάσιγκτον. Κατά τη γνώμη μου, οι συμφωνίες αυτές συνιστούν πρόοδο. Και θα ήθελα, κύριε Υπουργέ, να μας πείτε λίγα λόγια στο σημείο αυτό. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να συσφίξουμε τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ μας και ποιοι θα είναι οι τρόποι έμπρακτης εφαρμογής αυτής της συνεργασίας. Ευχαριστώ. Δεν είναι περίεργο που ζητούν πάρα πολλοί βουλευτέ το λόγο. Σα παρακαλώ λοιπόν όλους να σεβαστείτε το χρονοδιάγραμμα, δύο λεπτά, ούτω ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι. Ο κύριο Δία Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ ε, από πλευρά μου και την κυρία Ναπολιτάνο για την παρουσία της ενώπιον των δύο επιτροπών και της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Τονίζω και υπογραμμίζω και προσυπογράφω τα όσα ε, ανέφερε εισαγωγικά ο Πρόεδρος Λόπες Αγγιλάρ. Σύμφωνα απολύτως. Αν κοιτάξτε εσείς προς την Ανατολή και εμείς προς τη Δύση, θα συναντηθούμε στην ίδια θάλασσα. Μπορεί να σας φαίνεται αυτό μεταφορικό και λυρικό, αλλά είναι ουσιαστικό γιατί ε, είμαστε από τις δύο όχθες του Ατλαντικού, αλλά μας ενώνει ο Ατλαντικός συνεργασία. Δύο ζητήματα μας ανησυχούν. Ξέρω ότι το ένα δεν είναι της δικής σας αρμοδιότητας, αλλά ανησυχητικό παραμένει. Μιλώ για ε, το νόμο που μόλις ενέκρινε το Κογκρέσο για τα 10 δολάρια για κάθε Ευρωπαίο που μπαίνει στην επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών. Συμφωνείτε με την αμοιβαιότητα. 14 εκατομμύρια πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών κάθε χρόνο επισκέπτονται την επικράτεια της Ένωσης και είναι δημοκρατικός ο έλεγχος. Υπερισχύουν οι δημοκρατικοί στη στο Τώρα, σε ό,τι αφορά τη μετανάστευση, κάτι πιο θετικό. Ήσασταν χώρα υποδοχής μεταναστών, μεγάλη και σπουδαία, αλλά και η Ευρώπη. Εσείς έχετε δείξει ενδιαφέρον για την κοινοτική νομοθεσία και θα μπορούσαμε ενδεχομένω να θεσπίσουμε ένα ε, πλαίσιο συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα έτσι τόσο ευαίσθητα όπως είναι η διαχείριση των μεταναστευτικών ρευμάτων, το άσυλο, η ενσωμάτωση ε, των μεταναστών ή ε, ο έλεγχος των συνόρων. Ο συνάδελφος και φίλος μου Κάρλος ε, αναφέρθηκε στη θεώρηση διαβατηρίων με τρόπο έτσι κάπως επιφανειακό. Για εσείς γιατί δεν διαπραγματεύεστε με την Ευρώπη αλλά με κάθε κρατός μέλος χωριστά και τιμωρείτε χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Πολωνία κλπ. 16-20% των αιτήσεων θεωρήσεων απορρίπτονται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας αλλά και για την υπομονή σας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρκοπ. Uh, κυρία Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, εγώ ήμουν υπουργό μετανάστευση στο Ηνωμένο Βασίλειο και ο γιος μου, ο οποίος ζει στην Πιορία, στο Φίνιξ, στις Ηνωμένες Πολιτείες μου επιτρέπει να, τον, να επισκέπτομαι τη χώρα σας πολύ συχνά. Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω. Φυσικά ξέρω ότι οι ευθύνε σας αφορούν κυρίως τους ελέγχους και την ασφάλεια των πολιτών, τον είπα πάνω απ' όλα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που αφορά όλους μας που προσπαθούμε να ασχοληθούμε με θέματα όπως αντιτρομοκρατία. Και ποιο είναι αυτό, ότι πολύ εύκολα μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι κάποιες ομάδες, ε, κάποιες θρησκευτικέ ομάδες συνιστούν πρόβλημα. Και στην Ευρώπη και στην Αμερική αισθάνονται ότι είναι υποέλεγχο, ότι είναι ύποπτοι λόγω το, της συμπεριφοράς των εξτρεμιστών. Ε, μιλάω για τους α, μουσουλμανικούς πληθυσμούς που συνήθω ε, στη μεγάλη του πλειοψηφία είναι νομοταγεί πολίτε. αλλά δυστυχώς πληρώνουν το τίμημα τη ε, συμπεριφοράς των ε, εξτρεμιστών και των τζιχαντιστών. Δεν μιλάω μόνο για τους μουσουλμάνους μόνο. Το θέμα είναι πώς μπορούμε αποτελεσματικά να ανταλλάσσουμε προφορίες Ευρώπη και Αμερική που να μην τιμωρεί μεγάλου τομείς, μεγάλους πληθυσμούς, μεγάλες κοινότητες. Πώς μπορούμε να γίνουμε πιο επιλεκτικοί να αντιμετωπίσουμε δηλαδή αυτό το πολύ σοβαρό θέμα της αντιτρομοκρατίας. Thank you very much, uh, Ε, κύριε Λατφορτ, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ και εγώ με τους συναδέλφους μου και θέλω να ε, καλωσορίσω θερμά την Υπουργό. Εκτιμώ πάρα πολύ και ε, όπως και άλλοι τη σχέση μας στη Διατλαντική και τη συνεργασία για την ασφάλεια, αλλά για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη. Ε, πραγματικά αυτό μας απασχολεί πολύ στο Κοινοβούλιο, πέρα από πολιτικές ομάδες. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να σας ρωτήσω κάτι για το πώς βγαίνει κανείς ε, από τις Ηνωμένε Πολιτείες αφού τις έχει επισκεφτεί ξέρω ότι είναι δική σας απόφαση. Εσείς θα, ε, θα το αποφασίσετε όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Δεν ξέρω, ε, ίσως είναι θέμα κόστος ωφέλειας. Ξέρω, διαβάζουμε στον τύπο. Εάν τυχόν αποφασίσετε να μην δώσετε συνέχεια σε αυτό το θέμα, ενδεχομένω να υπάρχει δυνατότητα συζήτηση των συμπερασμάτων σας και συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή νομίζω του χρόνου θα σκεφτεί ένα τέτοιο σύστημα εισόδου-εξόδου ε, και θα πρέπει να το συζητήσουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να έχουμε κοινά ενδεχομένως συμπεράσματα ή να παρακολουθήσουμε τα συμπεράσματα και το υπόβαθρο. Και ένα δεύτερο, και έρχομαι τώρα στο σκέλος της δικαιοσύνης, άμα επιτρέπετε, Εξ όσων κατάλαβα, γιατί είμαι σε κάποια σύγχυση και θα πρέπει να το ομολογήσω, υπάρχει μια νομοθεσία που συνδέει το Visa Waiver, την ε, άρση της επιβολής ε, θεώρησης, με αυτή την υπόθεση της εισόδου-εξόδου από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είναι πέντε χώρες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ελπίζουμε σύντομα η μία να βγει από το, σύστημα, ε, τι θα γίνει ε, τελικά με τις αιτήσει που απορρίπτονται και ποια είναι η θέση του Κογκρέσου. Ευχαριστώ. Τελευταία ερώτηση για τον πρώτο γύρο, η κυρία Ρόπες. Ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω την κυρία Νεπολετάνο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αναφέρω κι εγώ κάτι που επισήμανε πρώτος ο κύριος Κίρκοπ. Το φαινόμενο της τρομοκρατίας, της διεθνούς τρομοκρατίας, τροποποίησε τις συνηθισμένες παραμέτρους αντιμετώπισης της τρομοκρατίας που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε μεμονωμένα οι διάφορες χώρες. κατά τη γνώμη μας, η τρομοκρατική ενέργεια κατά των δίδυμων πύργων τροποποίησε άρδιν τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην τρομοκρατία. Άρχισαν να χρησιμοποιούνται προληπτικά κάποια μέτρα, όπως έγινε και προληπτικά ο πόλεμος. Και η πρόληψη, αν δεν δίνει κάποια εχέγγυα, δημιουργεί πολλά προβλήματα. Ειδικά αν καταργεί κάποιες εγγύησεις. Το θέμα SWIFT είναι ένα από τα θέματα που εξετάσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά υπάρχουν και άλλα θέματα που κατοχυρώνουν την προστασία των δεδομένων. Από τη στιγμή που δεν έχουμε συγκεκριμένους στόχους και υιοθετούνται κάποια δυσανάλογα μέτρα, τα μέτρα αυτά είναι ορισμού αναποτελεσματικά. Ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι όπως ε, αυτοί που αναφέρθηκαν για τα προφίλ. Ίσως έτσι καταργηθούν κάποιες εγγύησεις και δεν ε, επιτυγχάνεται η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα. Η Ισπανία, όπως και άλλες χώρες, έχουν παράδοση στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Μπορεί όμως να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία με σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων και χωρίς ε, κατάργηση κάποιων ε, εγγύσεων. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμη και προληπτικά μέτρα, χωρίς όμως να χρησιμοποιούνται δυσανάλογα κάποιοι μέθοδοι που καταργούν εγγύησεις και ταυτόχρονα δεν είναι και αποτελεσματικές. Θα ήθελα ως προς το σημείο αυτό να έχουμε κάποια ανταλλαγή στο μέλλον. Καλώς, ολοκληρώσαμε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Υπουργό Ναπολιτάνο για να σχολιάσει τις παρατηρήσεις που ακούσαμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις ε, ερωτήσεις σας. Είναι πολύ σωστές, πολύ εστιασμένες. Θα ήθελα να ξεκινήσω με ένα πλαίσιο, να θέσω το πλαίσιο, ότι προσεγγίζουμε όλα τα θέματα με αμοιβαίο σεβασμό και στραμμένη στις κοινέ μας αξίες. Νομίζω προφανώς ότι πέρα από τις κοινέ αξίες έχουμε διαφορές, αλλά προσπαθούμε να τις ξεπεράσουμε. Σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα και τη διαφάνεια, η κυβέρνηση Ομπάμα θέτει ως βασική της προτεραιότητα τη διαφάνεια. Ελπίζω λοιπόν ότι αν υπήρξαν κάποια προβλήματα με την πρόσβαση στα επίσημα έγγραφα, πρόβλημα που αντιμετώπισε το Κοινοβούλιο, ελπίζω να επιληθεί. Πώς θα εφαρμόσουμε την αρχή αυτή. Είναι πολύ βασικό θέμα, γιατί πρέπει να περάσουμε από, την... από τις αρχές στη συμφωνία. Θα ήθελα να ακούσω και τις δικές σας ιδέες για το πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Αλλά πιστεύω ότι η κυβέρνηση Ομπάμα θα ήθελε να προχωρήσει όσο μπορεί πιο ταχαίω. Όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε ελέγξει τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε συζητήσει και νομίζω ότι υπάρχει μια, ένα καλό επίπεδο κατανόηση και αμοιβαία συνεννόησης για το τι πρέπει να γίνει. Θα περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν και τι δικέ σα συστάσει για το πώ θα περάσουμε από τις 16 αρχές σε μια πραγματική συμφωνία. Τώρα, για αυτό το νόμο το άστα των 10 δολαρίων συμπεριλήφθηκε στο νομοσχέδιο για τις πιστώσεις που πέρασε και από τα δύο σώματα της Βουλής. Και πιστεύω ότι ο Πρόεδρος θα υπογράψει αυτό το νόμο. Κοιτάξτε, αντίθετα από τι δικέ σα χώρε, κάποιες από τι δικές σας χώρες, εμείς δεν έχουμε μια ειδική υπηρεσία για να προωθήσουμε τα ταξίδια και τον τουρισμό. Ο στόχος λοιπόν του νόμου αυτού είναι να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα χρήματα για να βοηθήσουμε τους τουρίστες και τους ταξιδιώτες που θέλουν να επισκεφθούν τις ΗΠΑ. Δεν πάει στο γενικό κορβανά των Ηνωμένων Μπαίνει στην άκρη για να βοηθήσει την ανάπτυξη του τουρισμού να βοηθεί τους τουρίστες και τους ταξιδιώτες. Νομίζω λοιπόν ότι είναι και λογικός ο νόμος και σε αυτές τις δύσκολες μέρες σχνώνα η Ελλάδα με μειωμένους προϋπολογισμούς προσπαθούμε να χρηματοδοτήσουμε κάποια προγράμματα. Τώρα, για την αμοιβαιότητα και τα όσα είπατε σχετικά με αυτήν. Φυσικά πρέπει να σεβόμαστε την αμοιβαιότητα. Είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Τώρα για τη μετανάστευση. Θα ήθελα να σας μιλήσω όχι μόνο ως Υπουργός του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, αλλά και ως πρώην ε, κυβερνήτης μιας ε, μεγάλης συνοριακής πολιτείας της Αριζόνα, Έχω μεγάλη εμπειρία σε θέματα συνόρων και διαχείριση των συνόρων, γιατί μου και, και υπουργό δικαιοσύνη τη Αριζόνα, τη πολιτεία τη Αριζόνα. Νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε κάποιες καλές πρακτικές. Θα ήταν κάτι πολύ χρήσιμο και για τις δύο πλευρές. και θα ήθελα να συμμετάσχω στη, σε αυτή την ανταλλαγή ιδεών για αυτό το θέμα. Σε ό,τι αφορά το profiling. και κυρίως των ανθρώπων που ανήκουν σε συγκεκριμένες θρησκευτικέ ομάδες. Έχουμε συγκεκριμένους νόμους εναντίον τέτοιας διακριτικής μεταχείρισης, εναντίον αυτής της πρακτικής του profiling. Καθώς προσπαθούμε λοιπόν να εφαρμόσουμε τον νόμο, ε, δεν θα πρέπει να υποκύψουμε σε αυτή την πρακτική. Εδώ τώρα, σε σχέση με την ανταλλαγή δεδομένων για τους επιβάτες, έχουμε διαφορετικούς τρόπους για να εξετάζουμε αυτά τα δεδομένα. Ούτω ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος του profiling. Έχουμε, εστιάζουμε σε αυτούς που έχουμε προβληματικές πληροφορίες, αλλά αξιόπιστες και που δηλώνουν ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει κάποια σχέση με τρομοκρατικές οργανώσεις ή εγκληματικές οργανώσεις. Είναι πολύ σημαντικά αυτού του τύπου τα δεδομένα, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τους αλγόριθμους, τα δεδομένα, την τεχνολογία με σωστό τρόπο. Αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να ανοιγόμαστε προς τις διαφορετικές κοινότητες, ε, ιδίως όσες ε, αισθάνονται πολιορκημένες. Ε, λόγω ιδίω των δράσεων των εξτρεμιστών. Εμείς έχουμε μία διεύθυνση για τις αστικές και πολιτικές ελευθερίες. Η λειτουργία της είναι όχι μόνο να μην υποκύψουμε στο profiling, αλλά να μας επιτρέψει να ανοιχτούμε προς τις διάφορες κοινότητες, να τίνουμε χείρα βοηθείας για κοινότητες που μιλάω που είναι εγκαταστημένες φυσικά στις Πολιτείες. Σε σχέση με το θέμα της εξόδου μετά από επίσκεψη στις Ηνωμένε Πολιτείε, υπάρχει μια απόφαση που με περιμένει στο γραφείο μου και θα ληφθεί απόφαση μέχρι το τέλος του 2009. Μπορεί να μην ξέρετε κάτι, αλλά η νομοθεσία για την ε, παρέκκληση από την προϋπόθεση θεωρήσεων ε, αν δεν περάσει, δεν θα υπάρχει αυτή η περίπτωση παρέκκλησης. Το θέμα των ε, παρεκκλήσεων υποχρέωση θεωρήσεων ακούστηκε στι ερωτήσεις σας. Είσαστε μέλη του Κοινοβουλίου. Το θέμα των παρεκκλήσεων από την υποχρέωση θεωρήσεων είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό θέμα ε, και τμήμα των σχέσεων μεταξύ των διαφορετικών χωρών. πολλοί α, βουλευτές του Αμερικανικού Κογκρέσου δεν δέχονται αυτές τις παρεκκλήσεις. Γιατί είναι τμήμα του συστήματος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, επομένως, θεωρούν τουλάχιστον, θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στο πώς προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Υπάρχει πάντα η πιθανότητα το όλο πρόγραμμα να αμφισβητηθεί σε επίπεδο νομοθετικό. Και καταλαβαίνετε εσείς ε, ως βουλευτές ε, πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε σε αυτό το τομέα. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, δυσανάλογη απόκριση στην τρομοκρατία. Νομίζω ότι είναι ευθύνη μας να επιτύχουμε την ισορροπία και να καταλάβουμε ότι η ασφάλεια θα πρέπει να είναι εις βάρος της ε, ελευθερίας. Ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν πολύ σαφής στην ε, αρχική του ομιλία, όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του ως πρόεδρος, ότι δεν θα επιτύχουμε, δεν θα εξασφαλίσουμε την ασφάλεια ε, εις βάρος των αρχών που διέπουν τις ΗΠΑ και πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η δημιουργία αυτού του κράτους. Φυσικά θα πρέπει να κάνουμε αντικειμενική αξιολόγηση όλων των στοιχείων που έχουμε. Θα πρέπει να υπάρχει επικοινωνία, όπως σήμερα. Πρέπει να έχουμε μια σαφή προοπτική. Και θα πρέπει να χρησιμοποιούμε με σωστό τρόπο τις πληροφορίες που έχουμε για να προχωρήσουμε. Αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε και στο Υπουργείο Εσωτερική Ασφάλεια της ΗΠΑ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τις παρατηρήσεις και τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, μην ξεχνάτε το, τον περιορισμό που έχουμε με το χρόνο. Το πολύ δύο λεπτά παρακαλώ. Δεύτερος γύρος, ο συμπρόεδρος Μπροκ πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Στα αγγλικά. Εγώ θα σας παρακολουθήσω να μιλήσετε και λιγότερο από δύο λεπτά. Γιατί έχουμε δέκα ομιλητές παρακαλώ ακόμα. Και καλό θα ήταν να έχουν όλοι οι συνάδελφοι την ευκαιρία να πάρουν το λόγο. Θα ήταν ευγενικό αυτό. Παρακαλώ να κάνετε σύντομες ερωτήσεις και σχόλια. Η κυρία Χένις Πλάσχαρτ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ε, θα τα πω γρήγορα και ε, σύντομα. Σε ό,τι αφορά αυτό το ζήτημα των 10 δολαρίων Εκτιμώ αυτά που είπατε και καταλαβαίνω ότι έχει άλλες προτεραιότητες σήμερα η κυβέρνησή σας όπως είναι το σύστημα υγείας και τα λοιπά. Αλλά για μας είναι λίγο περίεργο να πούμε ότι προωθούμε τον τουρισμό και τα ταξίδια. Καλώς ορίσατε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ε, για να δώσετε τώρα φόρο 10 δολάρια με το καλημέρα σας. Ε, αυτό είναι κάπως περίεργο. Δεν θα είναι μόνο 10 δολάρια, θα καταλήξουμε στα 15-20 δολάρια. Λοιπόν, και η κατάσταση αυτή είναι περίεργη για μας, εν πάση Λοιπόν, επανέρχομαι σε αυτό που είπε η συνάδελφός μου η Βαρόνη Λάτφορτ για την ε, ε έξοδο χώρα και το πρόγραμμα κατάργησης υποχρέωσης θεώρησης διαβατήριο Visa Waiver στο νόμο αυτό συνδέεται με το στοιχείο της εξόδου και αδειμονώ να μάθω περισσότερες λεπτομέρειες ε, για τις πρόοδους που θα γίνουν τις επόμενες εβδομάδες. Είμαι βέβαιη ότι η συνάδελφος ε, είναι Βέλτ θα μιλήσει για το PNR. Το μόνο που θα ήθελα να τονίσω εγώ είναι μπορούμε σας παρακαλούμε να ε, ορίσουμε μία ημερομηνία για κοινή αναθεώρηση το συντομότερο. Ε, η συνθήκη της Λισαβόνας θα τεθεί σε ισχύ σύντομα και μια κοινή αναθεώρηση θα ήταν το ε, λιγότερο που θα μπορούσαμε να έχουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ε, καλωσορίσατε Καλώς ορίσατε στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη. Χαιρόμαστε που σας βλέπουμε ενώπιον μας. Ε, αυτό που κρατάμε είναι αυτό που μάθαμε από τον πρόεδρο Ομπάμα. Η καταπολέμηση δηλαδή της τρομοκρατίας είναι εξίσου σημαντική με την υπεράσπιση των ε, πολιτικών δικαιωμάτων. Δυστυχώς όμως αρχόμαστε να διαπιστώσουμε τώρα, συζητώντας με τους συνεργάτες σας, ε, ιδιαίτερα στο Υπουργείο σας για την εσωτερική ασφάλεια, αλλά και ορισμένους γερουσιαστές ε, ε, δημοκρατικούς, ότι τα μέτρα που προτείνονται ήδη εν μέρη είναι ακόμα πιο σκληρά και οξύτερα σε σχέση με εκείνα της προηγούμενης κυβέρνησης. Και για μας αυτό είναι κάτι το διχαστικό και μια δεχομένως διγλωσία που δεν μπορούμε να τη δεχτούμε ως κοινοβούλιο. Αυτό ισχύει και για το Visa Waiver και για τα 10 δολάρια. Παρακαλώ μας το εξηγήστε και για τις διαπραγματεύσεις για το SWIFT όπου θα πρέπει εμείς να επιμείνουμε ε, στις δικές μας, στις ευρωπαϊκές αξίες, ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων, ε, τα ευρωπαϊκά δικαιώματα των πολιτών θα πρέπει να μπαίνουν και αυτά και να εφαρμόζονται στις συμφωνίες με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας το διευκρινίσετε αυτό. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς εκτιμάτε το τρόπο που οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις συνεργάζονται με τις απόπειρες ε, του πρόεδρου Ομπάμα να κλείσει το Γουαντάναμο. Και όπως είπατε και εσείς, η διαφάνεια είναι σημαντική αξία της κυβέρνησης Ομπάμα. Και μάλιστα ο πρόεδρος Μπούς παραδέχτηκε την ύπαρξη μυστικών φυλακών. Γιατί δεν έχει ε, αποκαλυφθεί αυτό το σημείο. Δεν είναι μόνο το Γουαντάναμο που ήταν ε, ε, φανερή φυλακή, έχουμε και μυστικές φυλακές. Θα πρέπει λοιπόν, αποκαλύπτοντας ε, και την ύπαρξή τους ε, και την συνενοχή των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων με την κυβέρνηση Μπούς για τις παράνομες παραδόσεις, θα προκαλέσετε μεγαλύτερη συνεργασία από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για να συνεργαστούν μαζί σας και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Όχι επειδή πρόκειται για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά γιατί κάτι τέτοιο απαιτείται προκειμένου να είναι αποτελεσματικός ο κοινό αγώνας μας κατά της τρομοκρατίας. Για να μην δώσουμε κίνητρα ε, στους τρομοκράτες για στρατολόγηση νέων τρομοκρατών και για εκδίκηση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την παρουσία σας εδώ. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για θέματα που ενδιαφέρουν πολύ την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και για τις ελπίδες που έχουμε να αποθέσει στη κυβέρνηση Ομπάμα, δηλαδή επιστροφή στο κράτος δικαίου και στις ελευθερίες. Από την 11η Σεπτεμβρίου και κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπούς, αυτά, πώς να το πω, ήταν θέματα όπου κυριαρχούσε ο φόβος ή ο εκφοβισμός. Ε, αυτό ε, κυριαρχούσε στην πολιτική ασφαλεία. Ελήφθησαν πολλά μέτρα και κατά την άποψή μου τώρα είναι σημαντικό να έχουμε ανεξάρτητη αξιολόγηση των μέτρων και αποτίμηση και από κοινού με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή οι Ηνωμένε Πολιτείες να φροντίσουν να μην έχουμε μια κούρσα προς τα κάτω στα δικαιώματα των πολιτών ή στις προδιαγραφές για την ε, προστασία των δεδομένων, αλλά να είναι υψηλές οι προδιαγραφές και τα πρότυπα και να επιστρέψουμε και στην αρχή του απολύτου ε, κράτους δικαίου και τις βασικές ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να ξεφύγουμε από την προληπτική και γενική παρακολούθηση όλων των πολιτών, ανδρών και γυναικών. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και αισθητό. Γι' αυτό λέω χρειάζεται ένας απολογισμός και μία αξιολόγηση για να αποσυρθούν, να καταργηθούν μέτρα είτε δυσανάλογα είτε αναποτελεσματικά. Όλα αυτά λοιπόν είναι πραγματικά στο πνεύμα των κοινών κοινοτικών μας αρχών και των ελευθεριών. Χρειάζονται ορατές αλλαγές. Έχετε την υποστήριξή μας απολύτως σε αυτή την κατεύθυνση και έχω την αίσθηση ότι και στο Κογκρέσο αυτό συμβαίνει. Παρακαλώ συντομότερα προσπαθήστε. Κύριο Σταβάρες. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ. Πριν από ένα χρόνο ήμουν στο Σικάγο και δεν μπορούσα να ξεχάσω αυτό που είδα και τους πανηγυρισμούς για την εκλογή του Ομπάμα. Και πριν καν αποφασίσουν οι δημοκράτε ποιο είναι ο υποψήφιό του, εγώ ήξερα ότι έπρεπε να δώσω το παρόν στο Σικάγο εκείνη τη μέρα για να συμμετέχω κι εγώ στον εορτασμό για την εκλογή του Πρόεδρου Ομπάμα. Και παρόλο που είμαι από την αριστερή παράταξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εμεί ε, ε, βλέπουμε τον πιθανό αντιμερικανισμό μερικέ φορέ των Ευρωπαίων, αλλά με την νέα κυβέρνηση μεγαλύτερους δεσμούς φιλίας και μεγαλύτερο άνοιγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα υπάρξει ανταπόκριση και από την πλευρά των ε, Ευρωπαίων. Νομίζω ότι με τέτοιες ε, αγαστές σχέσεις ε, ο κόσμος θα ήταν ρόδινος. Έχω δύο θέματα που με απασχολούν όμως. Το πρώτο αφορά το Γουαντάναμο. Δεν ξέρω αν η κυβέρνηση Ομπάμα και αν οι ηγέτες ε, και των ευρωπαϊκών χωρών ε, πιστεύουν ότι 22 Ιανουαρίου θα είναι πραγματικά η επίσημη ημερομηνία κλεισίματος στο Γουαντάναμο γιατί κάτι τέτοιο θα δώσει αξιοπιστία σε όλες αυτές τις αποφάσεις και πολλοί πολίτες ε, του κόσμου περιμένουν αυτή τη χειρονομία από τον πρόεδρο Ομπάμα. Νομίζω ότι η ημερομηνία της 22ης Ιανουαρίου είναι συμβολική για μας, για όλο τον κόσμο και δεν θα πρέπει να πάει χαμένη για να μην, και να μην κλείσει το Γουαντάναμο. Ένας υπάλληλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκε σε μια πτήση για το Μεξικό που άλλαξε πορεία γιατί ε, βρισκόταν σε, έναν, σε έναν μαύρο κατάλογο επιβατών προ τι ΗΠΑ και μάλιστα για άγνωστου λόγου. Δεν καταφέραμε να εξακριβώσουμε γιατί. Υπάρχουν τέτοιοι κατάλογοι, μαύροι κατάλογοι επιβατών που δεν μπορούν να εισέλθουν στο έδαφο των Πολιτείων. Θέλουμε να μα ε, το σχολιάσετε. Η κυρία Στέλλα Νόκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας καλωσορίσω, κύριε Υπουργέ, Εκπροσωπώ ένα νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να μιλήσω για την ε, ανισότητα που υπάρχει μεταξύ των κρατών μελών της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για, την ε, θεώρηση, για τις θεωρήσεις. Είμαι Λετωνή. Κύριε Ναπολιτάνο, δεν νομίζετε ότι στο μέλλον οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχουν μια αμοιβαία συμφωνία για μια δυνατότητα ταξιδιών χωρίς θεωρήσεις. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αντιμετωπίζεται ως ολότητα, ως σύνολο στα πλαίσια αυτής της συνθήκης. Κυρία Ιντφελτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ, κυρία Ναπολιτάνο, μεγάλη χαρά σας βλέπω εδώ. Ο προκάτοχός σας είχε έρθει επίσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εκτιμήσαμε την παρουσία του, παρότι διαφωνήσαμε σχεδόν με όλα όσα μας είπε. Με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε. Ε, έχουμε σημειώσει μερικές θετικές εξελίξεις από τη νέα κυβέρνηση. Παρ' όλα αυτά, εξακολουθούν να παραμένουν κάποια μελανά σημεία, κάποιες ανησυχίες που ανέφεραν στην αδελφή μου. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ρωτήσω για τη συμφωνία για το PNR. Θα γνωρίζετε βεβαίω ε, ποια είναι η κατάσταση, ότι η συνθήκη τη Λισαβόνα θα τεθεί σε ισχύ ω ονούπο και ότι η συνθήκη δεν έχει ακόμα ακυρωθεί. Ίσως να βρεθούμε σε μια κατάσταση ε, όπου θα χρειαστεί να επαναδιαπραγματευτούμε. Πώς ε, αισθάνεστε για το περιορισμένο πεδίο. Πολλά είπαν για την, υπόθηκαν για την τρομοκρατία. Αλλά το PNR χρησιμοποιείται για μια πλειάδα στόχων που δεν έχουν καμία σχέση με την ε, τρομοκρατία. Ένα συναδελφό μου μίλησε για την κοινή αξιολόγηση τη αποτελεσματικότητα τη πολιτική αντιτρομοκρατία. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε κατεπηγόντω πληροφορίε για τα αποτελέσματα αυτή τη πολιτική. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι και στι ΗΠΑ και στην ε, Ευρώπη το πραγματικό πρόβλημα. Συγγνώμη, ποιο είναι το πρόβλημα. Να είστε πιο σύντομοι, παρακαλώ. Ε, έχω δύο λεφτά το ρολόι τρέχει. Θα τελειώσω λοιπόν τουλάχιστον την πρότασή μου. Επιτρέψτε μου να τελειώσω την πρότασή μου. Λοιπόν, το πρόβλημα ήταν πριν από τις 11 Σεπτεμβρίου, όχι ότι δεν είχαμε επαρκή δεδομένα για τους πολίτες, αλλά δεν υπήρχε επαρκής ε, συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των ε, υπηρεσιών και των χωρών. Ε, θεωρείτε ότι αυτό το πεδίο έχει βελτιωθεί, αυτό το μέτωπο. Ε, επίσης, ε, Πέρασα τις καλοκαιρινές μου διακοπές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασα πάρα πολύ καλά. Παρότι άφησα 10 δολάρια και 10 δακτυλικά αποτυπώματα, ελπίζω αυτό το μέτρο να μην συνεχιστεί. Ορίστε, 2.18 έγραψε το χρονόμετρο. Αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε και έτσι, αλλά στις 12 ακριβώς λήξεις και δεν θα έχει χρόνο να απαντήσει ο υπουργό. Γι' αυτό νομίζω καλό θα ήταν όλοι να τηρούν το χρόνο τους. Η κυρία Σινκλέρ. Καλώς ορίσατε, κυρία Υπουργέ, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι βέβαιη ότι στι ΗΠΑ πολιτείε έχετε μεγαλύτερη ελευθερία λόγου. Έχω εδώ τον μπρελόκ μου ε, που έλεγε κάτι που ε, είπε ο Ρίγκαν. Trust but verify. Να εμπιστεύεσαι, αλλά να επαληθεύεις κιόλα. Και αυτό κάνουμε κι εμείς. Έχω κάνει μια λίστα για το τι μας περιμένει την 1η Δεκεμβρίου. Μπορείτε να μας εγγυηθείτε ότι με μονομένες χώρες ε, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίζετε ξεχωριστά ως χώρα και όχι ως πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν πηγαίνουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς να θεωρούμαστε ε, ε, υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, όχι Ευρωπαίοι πολίτες. Και σε ό,τι αφορά τις αιτήσει, οι αιτήσει στο Λονδίνο είναι πολύ δύσκολο να περάσουν για να πάρουν βίζα χρειάζονται να ε, ε, δώσουν πάρα πολλά χρήματα. Uh, Σας ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα μία απάντηση σε μία συγκεκριμένη ερώτηση. Θα μπορούσαμε να στήσουμε μία μεικτή επιτροπή για την αξιολόγηση των καταχρήσεων θεμελιωδών δικαιωμάτων που διαπράχθησαν στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρώπη στο βωμό της καταπολέμησης της ε, τρομοκρατίας και ποια, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και το ρωτώ γιατί στην πατρίδα μου που είναι ε, χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μου μένει 1,5 λεπτό για να μιλήσω ακόμη, έχουμε 16 πολιτικούς κρατουμένους αυτή τη στιγμή, ε, φυλακισμένους της, αντιπολίτευσης ε, και ήδη ένα εξάμεινο εκτίουν ποινή με Κατηγορίε για συμμετοχή σε τρομοκρατικέ ενέργειε. Αυτοί οι άνθρωποι φυσικά είναι τελείω άσχετοι με την τρομοκρατία και η κράτησή του ε, συνιστά καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. απλώ προσπαθούν ε, να υψώσουν τη φωνή τους κατά των αδικιών που διαπράττονται στη χώρα μου και παρόλα αυτά βρίσκονται στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι με παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Και μάλιστα πολλές δυνάμεις ασφαλείας και αντιτρομοκρατική αστυνομία πηγαίνουν στις ε, κατοικίες των ανθρώπων αυτών και χωρίς ένταλμα, χωρίς ε, ε, δικονομικές εγγυήσεις, χωρίς μάρτυρες, κάνουν έρευνες στα σπίτια τους και καταπατούν και τα δικαιώματά τους ακόμη και στη φυλακή. Θα πρέπει και οι Αμερικανοί να πιέσουν τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, ώστε οι μετακομμουνιστικές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μην δακτυλοδεικνύουν τις Ηνωμένε Πολιτείες και να λένε αφού οι Ηνωμένε Πολιτείε το κάνουν, γιατί και εμεί να μην χρησιμοποιήσουμε στα ελληνιστικέ πρακτικέ κατά πάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων προκειμένου να υλοποιήσουμε του πολιτικού μα στόχου. Γιατί οι Αμερικανοί πολίτε ε, είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ήταν υπερήφανοι για την ελεύθερη χώρα του και τη δημοκρατικότητα. Θα πρέπει λοιπόν να πρωτοστατήσουν και πάλι στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κύριο Αλχαντράου, τελευταίος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώς ορίσατε κυρία μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι μέλος τη Επιτροπής Μεταφορών και έχω δύο ερωτήσεις που είναι σχετικές. Πρώτον, ε, φιλοδοξούμε να φτάσουμε σε ένα σύστημα λεγόμενο one-stop security. Τι σημαίνει αυτό. Ε, οι επιβάτες των αεροπλάνων να ελέγχονται μία φορά και όταν έχουν ε, ε, μια στάση σε ένα αεροδρόμιο για μετεπιβίβαση, transit, να μην ξαναελέγχονται. Αυτό βέβαια απαιτεί ε, συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, για να έχουμε μια κοινή στρατηγική ασφαλεία στα αεροδρόμια και μια κοινή προσέγγιση με κοινό χρονισμό για απαγορεύσεις υγρών και άλλα τέτοια. Εσείς συμμερίζεστε πρώτα απ' όλα αυτό το κοινό στόχο. Θέλετε να υπάρχει έλεγχος σε ένα και μόνο σημείο και πώς προτίθεστε να συνεργαστείτε με εμάς προς την κατεύθυνση αυτή. Το δεύτερο έχει να κάνει με τη μεταφορά ε, φορτίου, ε, κάργο. Ξέρετε ότι εγκρίθηκε ένας δόμος που λέει ότι ε, όλο το φορτίο που έρχεται, φτάνει σε λιμένες ε, των ΗΠΑ θα πρέπει 100% να ε, ελέγχεται με σκάνερς. Αυτό είναι και πάρα πολύ ακριβό, και πάρα πολύ άσκοπο. Εσείς θέλετε να το προωθήσετε αυτό, να το αποδυναμώσετε για να μην είναι αυτό εις βάρος και απειλή για το εμπόριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένων Πολιτειών και να μην έχουμε και πρόβλημα επιβολής του ιδίου μέτρου για φορτία και εμπορεύματα που έρχονται στην Ευρώπη από τι Ηνωμένε Πολιτείες. Χωρίς μικρόφωνο, Πρόεδρος. Κύριε Πρόεδρε, από την αρχή ήδη είχα ζητήσει το λόγο. Δεν είδα το όνομά στο κατάλογο, λυπούμε ειλικρινά. Κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Λυπούμε ειλικρινά, πραγματικά δεν είδα το όνομά στο κατάλογο. θα βάλω τα δυνατά μου και θα ανακεφαλαιώσω, θα συνοψίσω μάλλον τις απαντήσεις μου στις πολύ εύστοχες ερωτήσεις που διατυπώθηκαν και σε αυτό το γύρο. Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις μας και το πρόγραμμα σε ό,τι αφορά το σκέλος εξόδου από τις ΗΠΑ καθώς και τις εξαιρέσεις από τις ταξιδιωτικές θεωρήσεις. Θέλουμε όσο το δυνατό πιο στενή συνεργασία γίνεται και επαφέ, γιατί το θέμα αυτό έχει άμεσε επιπτώσει στη σχέση μας με τις ε, χώρες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά την ε, κοινή αναθεώρηση του PNR, ήδη έχει προγραμματιστεί μια τέτοια κοινή αναθεώρηση. Ήδη είχε προγραμματιστεί από πέρυσι μάλιστα. Και για πολλούς και διάφορους λόγους ακυρώθηκε αυτή η κοινή αναθεώρηση. Πάντως πολύ ευχαρίστως να οργανώσουμε μια τέτοια κοινή αναθεώρηση του PNR. Και πολύ ευχαρίστω να θέσουμε ήδη από σήμερα μια ημερομηνία για την πραγματοποίηση αυτής της αναθεώρησης. Πολύ ευχαρίστω. Χαίρομαι για αυτά που είπατε και πιστεύω ότι θα διευκρινιστούν πολλές σκέψεις για το PNR και πολλές προτάσεις για το πώς το εκλαμβάνονται πολλοί, ποιοι είναι οι περιορισμοί του. Και πιστεύω ότι έτσι θα διασκεδαστούν πολλές αμφιβολίες. Είμαι πρόθυμη να θέσουμε συγκεκριμένη ημερομηνία για κοινή αναθεώρηση του PNR. Ήδη από σήμερα. Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες και τον προβληματισμό του κ. Στράσε, για το κατά πόσο η κυβέρνηση Ομπάμα έχει αλλάξει στάση σε σχέση με την ε, κυβέρνηση Μπούς. Θα ήθελα να πω ότι ο πρόεδρος Ομπάμα ήταν ε, σαφέστατος και κατηγορηματικός. Θέλει ε, στενές σχέσεις ε, με τον ΟΗΕ και θέλει έναν ρόλο στις παγκόσμιες σχέσεις Αλλά ακόμη και αν στενιζόμαστε αυτέ τις αρχές, θα πρέπει να συνεργαστούμε σε συγκεκριμένα θέματα. Μερικά είναι εύκολα, όπω ο ορισμός μιας ημερομηνία και άλλα θέματα είναι πιο ακαθόδη. Εκεί θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειε μας. Θα ήθελα πάντως να τονίσω τη σημασία που έχει το SWIFT θα μπορούσαμε χάρη στο SWIFT ε, να διαλευκάνουμε θέματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Πιστεύω ότι η συζήτηση για το SWIFT είναι πολύ σημαντική για τη διεθνή ασφάλεια. Για την ασφάλεια όλων μας δηλαδή. Σε ό,τι αφορά τώρα το κλείσιμο του Γουαντάναμο, ο πρόεδρος έχει διατάξει να ολοκληρωθεί αυτό το κλείσιμο και μάλιστα γίνεται μια περιπτωσιολογική ανάλυση των διαφόρων υποθέσεων και το Γουαντάναμο περισσότερο χρησιμοποιήθηκε ως τρόπο συγκέντρωσης, ως συγκέντρωσης ε, και θα γίνει μια περιπτωσιολογική ανάλυση των υποθέσεων και θα κλείσουν οι συγκεκριμένες υποθέσεις των κρατουμένων. Το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνομιλίες ε, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες για την ε, ανάληψη πολλών κρατουμένων. Φυσικά ε, θα ολοκληρωθούν οι δίκες τους με βάση το αμερικανικό δίκαιο. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να περατωθεί. Είπατε ότι δεν θα πρέπει να γίνει ισοπαίδωση ή ευθυγράμμιση με τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή σε ό,τι αφορά τι πολιτικέ ελευθερίε και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Αλλά δεν νομίζω ότι γίνεται μια τέτοια υποβάθμιση ή εξίσωση προ τα κάτω. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια ασφάλεια που δεν θα είναι δυσανάλογη με τον κίνδυνο. Προσπαθούμε να ελεγχιστοποιήσουμε τους κινδύνους και ταυτόχρονα σεβόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πολιτικές ελευθερίες. Αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερα προσφυλές στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και σε εσά. Πολλοί, σας αναφερθήκα, πολλοί από σας αναφερθήκατε στην ε, κατάργηση των αναποτελεσματικών μέτρων και είπατε ότι ορισμένα από τα μέτρα αυτά είναι περιτά. Μα σίγουρα κανείς δεν θέλει να εφαρμόζει αναποτελεσματικά μέτρα αλλά μερικές φορές είναι πολύ δύσκολο να καταμετρηθεί μία αρνητική επίπτωση ή μία έλλειψη αποτελεσματικότητας. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα που γνωρίζαμε, θα το αντιμετωπίζαμε. Και δεν ξέρουμε σε ποιο βαθμό ορισμένα μέτρα είναι αποτελεσματικά, αναποτελεσματικά. Ή τι πρέπει να κάνουν οι επιβάτες πριν ε, επιβιβαστούν, για παράδειγμα, στην πτήση τους. Εμείς θέλουμε να αποτρέψουμε αρνητικές ενέργειες Γι' αυτό και θεσπίσαμε αυτά τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα του αεροπλάνου που άλλαξε πορεία, θα ήθελα να σας πω ότι εξετάστηκε ε, αυτή, αυτό το μέτρο και νομίζω ότι ήταν σωστή αυτή η αλλαγή πορείας. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο προς το παρόν. Σε ό,τι αφορά πάλι την εξαίρεση από τι θεωρήσεις, που ισχύει για ορισμένε μόνο ευρωπαϊκέ χώρε και όχι για άλλε. πέρυσι ε, προσθέθηκε αυτή η άρση των θεωρήσεων για άλλε 7 χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά η νομοθεσία μα ε, επιβάλλει η άρση αυτή να γίνεται περιπτωσιολογικά αναχώρα μετά από συγκεκριμένη αξιολόγηση. Δεν μπορεί να γίνει συλλήφθη για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τη χρήση τη συμφωνία PNR και αν θα πρέπει να γίνει αναδιαπραγμάτευση γιατί τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για κατάλληλου σκοπούς. Θα ήθελα να σας πω ότι με βάση τη συμφωνία τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για να εξακριβωθεί τρομοκρατία ή σοβαρό διεθνές έγκλημα. Μόνο για αυτούς τους σκοπούς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία PNR. Και Δεσμευόμαστε από τη συμφωνία αυτή. Αλλά όπως είπα και προηγουμένως, θα πρέπει να γίνει μια αναθεώρηση της συμφωνίας PNR και μάλιστα από κοινού. Η Ευρωβουλευτής Σενκλέρ Είπε κανεί ότι όταν ε, φτάνει στι Ηνωμένε Πολιτείε και επισκέφτεται τι Ηνωμένε Πολιτείε δεν θα πρέπει να χάνει την εθνική του ταυτότητα. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο. Πραγματικά δεν το φοβάμαι αυτό. Σε ό,τι αφορά την ε, επαχθή εφαρμογή του συστήματος θεωρήσεων και την υπερβολικά δαπανηρή εφαρμογή της, εμείς θέλουμε ταξιδιωτικές ανταλλαγές, ε, τουρισμό. Θέλουμε όλο και περισσότεροι πολίτες να έρχονται στις ΗΠΑ και να έχουν μια προσωπική εμπειρία όπως είχατε εσείς στο Σικάγο. Έτσι θα αρθούν τα πέπλα του μυστηρίου και θα καταρριφθούν κάποιες θεωρίες που εμφανίστηκαν για τις ΗΠΑ. Πολιτείε. Οπότε αυτά τα μηνύματα θα τα διαβιβάσω στο αρμόδιο Υπουργείο που είναι το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε ό,τι αφορά το One Stop Security για τα αεροπορικά ταξίδια, πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η πρόταση. και πραγματικά θα μπορούσαμε να εμπνευστούμε από αυτή. Δεν ξέρω αν βραχυπρόθεσμα είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, πάντως ενδιαφέρουσα πρόταση για να διευκολυνθεί η μετακίνηση. θα το σκεφτώ περαιτέρω. Σε ό,τι αφορά την ανάγκη με, ε, σάρωσης, screening στο σύνολο των φορτίων των εμπορευμάτων. Πραγματικά είναι εξαιρετικά δαπανηρή αυτή η διαδικασία και χρονοβόρα και είπα το επίσημα στο Κογκρέσο και έχω και επιχειρήματα που το δεκμηριώνουν. Γι' αυτό και θέλουμε να αναθεωρήσουμε αυτό το μέτρο για να γίνεται πλήρης θάρρωση όλων των εμπορευμάτων. Αυτό το μέτρο θα πρέπει να επικεντρωθεί στους κινδύνους και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ελεγχιστοποιήσουμε τον κίνδυνο. Βέβαια, έχουμε επίγνωση ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο. Δεν ζούμε σε αποστηρωμένο περιβάλλον. Πάντως πολλά από τα μέτρα που ε, εξετάσαμε σήμερα, όπως και το screening του φορτίου, ε, προσπαθούν να υλοποιήσουν αυτό το στόχο. Σας ευχαριστώ και για την εισαγωγή σας κύριε Υπουργέ και για τις απαντήσεις της ερωτήσεις σας. Ήρθατε σε μια σημαντική εβδομάδα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί αυτή τη εβδομάδα αποφασίστηκε να κυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας και τίθεται πλέον σε ισχύ την 1η Δεκεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι αρμοδιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι εσωτερικέ υποθέσει. και επομένω έχει νόημα να συναντηθούμε εδώ. Οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι πρόδρομο σε αυτά τα θέματα. Σας ευχαριστώ λοιπόν που ήρθατε και συμφωνούμε ότι πρέπει να βρούμε ισορροπία μεταξύ προσωπική ελευθερία και ασφάλειας. Εδώ βεβαίω μπορούμε να έχουμε διαφορετικές απόψεις, εμείς και εσείς. Αλλά και εμείς στο εσωτερικό μας έχουμε πολλές απόψεις, ε, όπως και εσείς στο δικό σα το Κογκρέσο. Είναι ανάλογη η κατάσταση. Νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί η σωστή ισορροπία και να εξασφαλιστεί ότι οι εχθροί της ελευθερίας δεν θα κάνουν ό,τι θέλουν γιατί το παρακάνουμε με τα μέτρα ασφάλειας. Πρέπει να υπρασπιστούμε και τα δύο μέτωπα, ασφάλεια και ελευθερία. Πριν από δύο-τρία χρόνια επισκέφθηκα τον Γκουαντάναμο και ξέρω πολύ καλά γιατί μιλάω. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να δούμε και την οικονομική διάσταση του θέματος. Ε, σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε για την σάρωση, για το σκάνι. Θα πρέπει επίση ε, το μέτρο αυτό να έχει και μία να ληφθεί υπόψη την οικονομική του διάσταση. Θα πρέπει να είναι εύλογο. Ε, δεν θα πρέπει να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο εμπόριο και στις θέσεις απασχόλησης. Με την νέα συνθήκη της Λισαβόνας θα πρέπει οι Ηνωμένε Πολιτείε να αντιμετωπίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο, ιδίως ό,τι αφορά την άση των θεωρήσεων. Και ο πρόεδρος Ομπάμα, η κυβέρνηση συνολικά Ομπάμα και το Υπουργείο Ιστορικής Ασφάλειας βράται διαφορετικά από ό,τι προηγούμενη κυβέρνηση. Όπου οι πολιτικές της δεν οδήγησαν σε θετικές εξέλιξεις για κανένα. Πάντως δεν είναι θέμα μόνο της κυβέρνησης αυτό και όλα τα προηγούμενα. Έχει σημασία και η άποψη του Κογκρέσου. Ε, έχει σημασία ο διατλαντικός διάλογος, οι επαφές μεταξύ των αρμοδίων επιτροπών. Θα πρέπει να γίνουν συζητήσεις και σε αυτό επίπεδο. Και βεβαίως και σε επίπεδο κυβερνήσεων, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια κοινή άποψη, σε κοινέ απόψεις. Νομίζω ότι ένα σεμινάριο για την άρση των θεωρήσεων πούμε, και την προστασία των δεδομένων θα μπορούσε μια καλή ιδέα για να φτάσουμε σε αυτές τις κοινέ απόψεις. Και ελπίζουμε ότι οι εισηγητές του Κοινοβουλίου θα έχουν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις απόψεις τους στις Ηνωμένε Πολιτείε για τα θέματα εσωτερικών, για τα οικονομικά θέματα, για την ε, οικονομική νομοθεσία του G20 που δεν θα πρέπει να πηγαίνουν στην λάθος κατεύθυνση γιατί αν συμβεί κάτι τέτοιο όλοι θα πληρώσουμε το κόστος. Ε, σας ευχαριστώ κύριε Υπουργέ που μας δώσετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για όλα αυτά τα θέματα.